Vamos a continuar la sesión por lo que... Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρακαλώ ή να καθίσετε ή να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη αφορά τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόφαση της 15ης Ιουλίου σχετικά με την θερινή δέσμη για την ενέργεια. Ο κύριος Εύκοβιτς έχει το λόγο.